η διαστολή με το πώς που καλύπτεται από, τους, ε, ε, από τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, είναι όλες οι πράξεις γενικής εφαρμογής, δηλαδή δεν μπορούν να προκύψουν μεμονωμένες κατά περίπτωση αποφάσεις και δεν περιέχουν ουσιαστικά στοιχεία που τροποποιούν το, τη βασική νομοθετική πράξη διότι προσθέτουν νέες υποχρεώσεις, ε, δηλαδή να αλλάζουν το πνεύμα αν θέλετε, απλώς υπησαρχόμαστε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή και αυτός είναι και ο στόχος των δύο πράξεων διότι όλες αυτές ε, οι διατάξεις ε, είχαν κρυθεί υπερβολικά τεχνικές ε, για να ρυθμιστούν στο βασικό κανονισμό και ως εκ τούτου τα τρία θεσμικά όργανα συναποφάσισαν ότι θα συμπεριληφθούν σε ένα τεχνικότερο, σε μια τεχνικότερη πράξη που θα συζητηθεί και σε τεχνικό επίπεδο. Οι υποχρεώσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ε, κατεξουσιοδότηση πράξει διαφέρουν σε σχέση με τι εκτελεστικέ πράξει. Ε, δεν υπάρχει καμία επιτροπολογία, δεν ψηφίζουν τα κράτη-μέλη. Αντίθετα, χρειάζεται, ε, υπάρχει υποχρέωση μάλλον διαβούλευση όλων των εμπειρογνωμών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, αυτό έγινε. Είχαμε πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Το, εξηγώ, το εξηγούμε στον ε, ε, επεξηγηματικό συγγνώμη, σημείωμα και είχαμε σε αυτές τις πέντε ομάδες εθνικούς εμπειρογνώμονες και από τα συνδεμένα με το Σέγγεν κράτη και από το Κοινοβούλιο. Είχαμε από τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ παραδείγματος χάρη εμπειρογνώμονες που παρήθαν σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα. Δυστυχώ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία το 2013, δεν είχαμε την ε, νομική βάση που, είχαμε, που χρειαζόμασταν. Νομίζουμε τώρα ότι μπορούμε να συζητήσουμε για την εφαρμογή των διατάξεων για τα ταμεία για να αρχίσουν να τρέχουν όλα κατά τη διάρκεια του 2014. Αυτό τουλάχιστον ευελπιστούμε τότε δεν ήταν ξεκάθαρο αν όλες αυτές οι διατάξεις θα συμπεριλαμβανόντουσαν σε εκτελεστική ή σε κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, είχαμε συμπεριλάβει αυτές τις διατάξεις σε δελτία ε, και είχαμε 78 ε, ερωτήσεις. Ε, είχαμε βάλει σε ένα πίνακα ερωταπαντήσεων και συζητήθηκαν αυτά τον Οκτώβριο του 2013 στη δεύτερη σύσκεψη των εμπειρογνωμών, Στην τρίτη που έγινε το Φεβρουάριο του 2014 τότε είχαμε ήδη την πολιτική συμφωνία επί των ταμείων και μπορέσαμε να καταθέσουμε ένα ακέραιο κείμενο. Στις 4 Απριλίου έγινε η τέταρτη συνεδρία των εμπειρογνωμόνων και πάλι πριν εγκριθούν επίσημα οι κατεξουδότηση πράξη και στις 6 Ιουνίου μια τελευταία σύσκεψη μετά την ε, διεπηρεσιακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χτενή στο κείμενο νομική υπηρεσία και το καθεξής και μπορέσαμε στις 6 Ιουνίου να το παρουσιάσουμε, παρουσιάσουμε την τελευταία εκδοχή των εμπειρογνωμόνων μετά από αυτό δεν λάβαμε πλέον ερωτήσεις από κανέναν. Η πρώτη ε, πράξη για ε, τις ε, αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου ε, ε, ε, περιέχει τους κανόνες σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν για την εφαρμογή των διατάξεων στα ταμεία τα κράτη-μέλη είναι κέρια σημασία σε η πράξη, διότι προτού αρχίσουν να χρησιμοποιούν το ταμείο τα κράτη-μέλη, χρειάζονται μια ε, ειδικώ ε, διορισμένη για αυτό το σκοπό ε, αρχή, αρμόδια εθνική αρχή. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί φυσικά η αρχική πράξη. Αν δεν εγκριθεί αυτή η Η πράξη, είναι απαραίτητο να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν. Ε, όντως τα κράτη-μέλη ε, ήδη εργάζονται, ξέρουν ότι συνεχίζονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν είναι και τόσο καινούργια ε, οι κανόνες εξάλλου. Και δεν είναι περίπλοκοι διότι προκύπτουν από τα ταμεία όπως θα ξέρουμε. Το Solid Funds εναρμονίζει τη λειτουργία και των διαρθρωτικών ταμείων. Ε, λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσει του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι ναι ε, νέο το περιβάλλον, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε για σωστή εφαρμογή είναι σταθεροί κανόνες. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ευκολότερα να ελέγξει την δραστηριότητα των κρατών μέλων. Δεν γίνεται αυτό χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ε, ε, υπάρχει η περίοδος παρατήρησης ε, και ελέγχου. Έχουμε αρχίσει έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβρη και βλέπουμε ότι ακόμη δεν μπόρεσαν να εγκριθούν ε, εθνικά ε, προγράμματα και απευχόμεθα μια περαιτέρω καθυστέρηση αν δεν ε, συντρέχει κάποιος βάσιμος λόγος. Θα σας παρουσιάσω τώρα το περιεχόμενο της κατεξουσιοδότησης αυτής της πράξης. The first act and then my colleague Έχουμε την πρώτη πράξη, η συνάδελφος θα επεξηγήσει τη δεύτερη. Περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, καταρχήν γενικές διατάξεις με τους ορισμούς και τα δύο κεφάλαια, το 2 και το 3 που είναι ζωτική σημασίας και αφορούν τα ζητήματα που απασχολούν τις αρμόδιες αρχές, το τμήμα υπαριθμών 1 ε, μιλά για το πώς ορίζεται η αρχή αυτή από το κράτος μέλος και πώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο διορισμός ή να αποσυρθεί ε, αν η αρμόδια αρχή δεν δρά καταλήλως. Το δεύτερο τμήμα ε, ορίζει το τι θα κάνει η αρμόδια αρχή ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία Δηλαδή, τι θα γίνει εάν υπάρξει εξωτερική ανάθεση ή εξουσιοδότηση σε τρίτους και στη συνέχεια τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής ως προς τις δημόσιες παρεμβάσεις, δηλαδή πώς γίνονται επιδοτήσεις και ούτω καθεξής και σε αυτή την περίπτωση οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν μία ανοιχτή διαδικασία και να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τις ελεγκτικές αρχές, πώς θα ε, ελέγξουν την αρμόδια αρχή και θα ε, αναφερθούν στην Επιτροπή εάν ε, υπάρχουν προβλήματα. Και το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τις τελικές διατάξεις, είναι πολύ απλό. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες αυτών των κεφαλαίων ή της πράξης. Θα θέλαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία παρατήρησης να σας επεξηγήσω αν θέλετε γιατί και από πού προέρχονται αυτές οι διατάξεις και η Στέφανη Χάρδη θα σας μιλήσει για την πράξη που αφορά την ε, πληροφόρηση και την ε, δημοσιοποίηση. Όπως σας είπα, αυτή η κατεξιδότηση πράξη αποτελεί ένα συμπλήρωμα της νομικής βάσης που είναι απότοκη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έτσι ώστε να ε, λάβουμε υπόψη το άρθρο 53 του κανονισμού και να πληροφορούμε το κοινό. Υπάρχει και μία εφαρμοστική πράξη σε σχέση με τις ε, μπλε σημεούλες και ούτω καθεξής, blue flags. Όπως ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, η χρήση των ε, κοινοτικών, των ευρωπαϊκών ταμείων και γι' αυτό ορίζουμε τα προαπαιτούμενα ώστε τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν το κοινό και τους δικαιούχους. Πρόκειται για υποχρεώσεις των κρατών μελών. Οι κανόνες θα συζητηθούν, μάλλον συζητήθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 και τον Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2014 με την ομάδα εμπειρονομών και στις 6 στις 6 Ιουλίου πήραν τελική μορφή με βάση ε, τις αποφάσεις για το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και στο τέλος του μήνα του Ιουνίου παρουσιάστηκαν το, στο Κοινοβούλιο. Ορίσαμε και τον χρηματοδοτικό κανονισμό, τους ίδιους τους κανονισμούς, καθώς και τον οριζόντιο κανονισμό για τα διαρθρωτικά και χρηματοδοτικά ταμεία. Θα πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη το μέγεθος και τη φύση των ταμείων Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα για να μην υπάρχει υπερβολικό άχθος με διοικητικού περιεχομένου πράξης. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη και οι δικαιούχοι μπορούν να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν ε, τις ε, λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει φυσικά να υπάρχει ίση μεταχείριση πάλι. Σε σχέση με τη φύση των ταμείων υπάρχουν ορισμένα ε, ευαίσθητα σημεία. Υπάρχει ο εμπιστευτικός χαρακτήρας που επιτρέπεται και για να υπάρχει και προστασία προσωπικών δεδομένων πρωτίστως αλλά μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ε, λαμβάνουμε υπόψη τέσσερις ε, συνιστώσεις ή υποχρεώσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διαδώσουν και με όλα τα μέσα τα βασικά στοιχεία που διέπουν τα ταμεία με βάση τα εθνικά προγράμματα. Επίσης, στη συνέχεια υπάρχει υποχρέωση προς τους δικαιούχους ή οποιαδήποτε φορέα που λαμβάνει ε, χρήματα να το γνωστοποιήσει ε, γραπτός με όλα τα μέσα έτσι ώστε να γνωστοποιήσει πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια. Στο τρίτο τμήμα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν όλους τους ενδυνάμει δικαιούχους για το πώς αυτά τα κονδύλια μπορούν να ε, ληφθούν έτσι ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους τους δικαιούχους. Τέλος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κατανοήσουν τα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να υπάρχει δημοσιοποίηση στοιχείων μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας. Θα ήθελα, λέει η Πρόεδρος, να τελειώσετε με την παρουσίαση για να μπορέσουν και οι βουλευτές να λάβουν το λόγο. Ναι, εντάξει, τελείωσε. Uh, λοιπόν, η κυρία Βίξτρομ ε, πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληροφόρηση αυτή που ήταν απαραίτητη άλλωστε. Και οι δύο ε, κατεξουδότηση πράξεις ε, παρουσιάστηκαν, κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο τέλη Ιουλίου και αυτόματα τίθεται σε ισχύ ε, η νομοθεσία. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και πλήρης αξιολόγηση διότι είναι και η πρώτη φορά που λαμβάνουμε τέτοιου είδους κατεξουδότηση συγγνώμη, πράξη στην Επιτροπή μας η Κομισιόν τώρα βιάζεται ότι είναι τεχνικό το θέμα και να ξεμπερδεύουμε. Ξέρουμε όμως πάντα ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε εδώ για να αξιολογούμε οτιδήποτε κατατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ επιμένω το άρθρο 105 του κανονισμού να ε, ε, εφαρμοστεί πλήρως. Ε, ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και τις δύο παρουσιάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανονισμούς και τις κατεξοδότηση πράξης. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μεν εξαντλητική και εκτενής η ε, ε, εξήγηση, αλλά εξίσου συγκεχημένη και σκοτεινή για μένα. Έχει σημασία όμως και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας το εξής. Είναι κοινό μυστικό ότι δεν συμφωνήσαμε τα θεσμικά όργανα για την ε, εφαρμογή των κατεξοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών. Και θέλω να σας θυμίσω γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να μην το γνωρίζετε, όταν ε, διετέλεσα εισηγητής για ε, τον κανονισμό 539 κάθετος 2001 ε, για τις θεωρήσεις στην κοινότητα διαβατηρίων. Μετά από μια πολύ εντατική νομοθετική προσπάθεια ετών, Υπήρχαν βασικές συμφωνίες επί της αρχής με όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά διαφωνήσαμε και συγκρουστήκαμε μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή χρήση σε μια κοινή επικεφαλίδα των κατεξουδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ε, ήταν δεδομένη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο δικαστήριο κατά του Κοινοβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που ακόμα ε, είναι υπό τη δική της δικαιοδοσία ε, του δικαστηρίου μάλλον. Αλλά άκουσα να αναφέρεται ο κανονισμός για το Ταμείο Σύλλου και Μετανάστευσης και επιλέξει είπατε ότι επιπλέον ο κανονισμός αυτός έρχεται να συμπληρωθεί από μία εκτελεστική πράξη. Για να μου το εξηγήσετε αυτό παρακαλώ. Και θα ζητήσω από τον Αντουάν που ξέρει τα θέματα αυτά σε βάθος, τα τεχνικά, να μου εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Κατεδίαν, όχι τώρα. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στο δικαστήριο για τις καταξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις όταν το Κοινοβούλιο προβάλλει την άποψή του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διατρανώνει, τώρα μας λένε ότι είναι το ίδιο. Ε, για τον ίδιο κανονισμό, κάτι εξοδότηση και εκτελεστική πράξη. Αυτό είναι το σχόλιο μου, αλλά και αυτό χρόνο και η αγωνία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, ευχαριστώ, κύριε Δίας Δεμέρα. Είμαι βέβαιος ότι η γραμματεία θα σας διαφωτίσει ε, δεόντως και διμερός στη συνέχεια. Άλλο συνάδελφο θέλει το λόγο, παρακαλώ. Γνωρίζετε ότι οι συντονιστές συζήτησαν ε, το πρωί αυτό το θέμα και θα επανέλθουν ε, για να αποφασίσουν στην επόμενη συνεδρίασή τους για να δούμε πώς θα χειριστούμε όλα αυτά τα θέματα. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο τώρα να προσθέσει τίποτα να ρωτήσει. Θέλει μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλος, να σας ευχαριστήσω όλους για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας, στην ημερήσια διάταξη. Που είναι η έκθεση 2010-2014 ε, για την τελική έκθεση εφαρμογής. Ο κύριος Λούιτσι Σορέκα είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Είναι Διευθυντής Εσωτερικής Ασφάλειας. Παρακαλείτε να μας παρουσιάσει αυτή τη τελική έκθεση εφαρμογής στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Θα επανέλθουν οι, οι συντονιστές συγγνώμη, για να το ξανασυζητήσουν. Παρακαλώ κύριε Σορέκα. Δεν τον βλέπω όμως. Παρακαλώ. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Είμαι Διευθυντής Αρμόδιος για την Ιστορική Ασφάλεια στη Γενική Διεύθυνση HOME. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα σε όλα τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Ελευθεριών την τελική εκθεση εφαρμογη εφαρμογή στρατηγικής εσωτερική ασφάλειας 2010-2014 είναι μια ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. Θυμούμε ότι ε, πέρυσι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ε, μια νέα εσωτερική ασφάλεια, μια στρατηγική δηλαδή, για την περίοδο 2015-2020 και συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο το ζήτησε αυτό στο ψήφισμά του 2636. Επί τη βάση αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης την πρωτοβουλία στην ανακοίνωσή της να βασιστεί στις ενδείξεις του και υποδείξεις του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα αυτό. Επίσης θα γνωρίζετε ότι το ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό, μια ενημέρωση ε, της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια τι λεγόμενες στρατηγικές κατευθυντήριες ε, γραμμές του Ιουνίου 2014. Έξω και η εκθεσή μας λοιπόν ε, που έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Ε, κάνει μια ανασκόπηση την περασμένη πέντα ετία, αλλά παρουσιάζει και τις προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον για να ξεκινήσει μια συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, τον ιδιωτικό τομέα, τα πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών και θα σας εξηγήσω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οργανώνει αυτή τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου καταρχάς και πάρα πολύ σύντομα να κάνω μια αναφορά ε, στο παρελθόν, στην ανασκόπηση λοιπόν ε, της περασμένης περίοδου και τα επιτεύγματά μας, γιατί και αυτό θα μας βοηθήσει να θέσουμε τα ορόσημα και τις βάσεις για την επόμενη στρατηγική δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την έκθεση, ε, καταλήγει ε, λέγοντας ότι σε νομοθετικό και επιχειρησιακό επίπεδο και η Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τα μέσα τους για να προστατεύουν καλύτερα ε, την κοινωνία, την οικονομία και τα δικαιώματα των πολιτών για καλύτερη και πιο στενή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής της τάξης και αυτό βέβαια έχει ήδη γίνει και σε επιχειρησιακό επίπεδο και έχει φέρει αποτελέσματα σε ε, αστυνομικές έρευνες διασυνοριακές και ένα μεγάλο επίτευγμα ήταν πολιτική κατά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και αυτά τα έχει αναλάβει η Europol και η Eurojust, το Frontex και η Olaf. Οι δυνατότητες που υπάρχουν έχουν επίσης ενισχυθεί, καθώς επίσης και ενισχύθηκε η εκπαίδευση στη ΣΕΠΟΛ, την Αστυνομική Ακαδημία, ε, αλλά και το ε, νέο SIS-2 και το Euroson. Μια νέα νομοθεσία στρατηγική προωθήθηκε το 2010 με 2014 για την καταπολέμηση του τράφικινγκ, για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, χώρο, στη θάλασσα και ε, ένας νέος μηχανισμός για την προστασία ε, των θυμάτων ε, στο αστικό δίκαιο και άλλα. Βάσει όλων αυτών λοιπόν και βάσει και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου άρχισε μια διαδικασία διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αφορά το δεύτερο τμήμα τώρα, το δεύτερο μέρος της έκθεσης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό είναι τώρα το περιεχόμενο του δεύτερου μέρους της ε, έκθεσης, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη συνέχεια και την αλλαγή. Ε, όταν ανανεώνουμε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να ενισχύσουμε και να δυναμώσουμε ε, ό,τι λειτουργεί σωστά και να αλλάξουμε τα κακό κείμενα ή εκείνα που δεν αποδίδουν όσο θα θέλαμε. Από τη μια λοιπόν συνεχίζουμε την εφαρμογή με την ε, υλοποίηση της νομοθεσίας και ε, εδραίωση των ε, όσων έχουμε πετύχει και με περισσότερη πρακτική συνεργασία και ενισχυμένη. Από την άλλη όμως πρέπει να βρούμε, πώς να το πω, ένα νέο αφήγημα για να μπορεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει και την κοινωνία και τα δικαιώματα των πολιτών. Έτσι λοιπόν η νέα στρατηγική θα αναθεωρήσει τη δράση αυτή για να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, νέες απειλές, διατηρώντας ταυτόχρονα τους πέντε στρατηγικούς στόχους ε, της σημερινής στρατηγικής. Διότι αυτοί οι πέντε στόχοι καλύπτουν όλοι τις βασικές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να σας θυμίσω αυτό. Ε, ε, η καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας, ε, της ριζοσπαστικοποίησης, της στρατολόγησης, αύξηση της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο για πολίτες και επιχειρήσεις, ενίσχυση της ασφάλειας, διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών και θεομηνιών. Αυτοί οι πέντε στόχοι χρειάζονται να παρουσιάζονται τώρα με ένα νέο τρόπο, με μια νέα αφήγηση όπως λέμε. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βασιστεί σε τέσσερις πυλώνες που στα αγγλικά είναι τα αρχικά P και 3I. Το P είναι protection, προστασία και τα 3I είναι information, innovation και international cooperation, δηλαδή ενημέρωση, καινοτομία και διεθνής συνεργασία. και θα πρέπει πάντα η προσέγγιση μας να έχει στο κέντρο της τον πολίτη. Αυτό θα πρέπει να είναι ο γνώμονας και η πηξίδα μας στη νέα στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια. Θα πρέπει νομίζουμε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να ε, εμπεριέχονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη νέα στρατηγική για να υπάρχει και υποστήριξη από το λαό για τις δράσεις μας. για να πετύχουμε ένα αμοιβαίο όφελος. Επίσης θα πρέπει να βρούμε ε, καλύτερη νομική βάση ε, και αηφορία βιωσιμότητα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν και γι' αυτό το σκοπό ήδη έχουμε ε, αρχίσει μια νέα συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων που έτσι κι αλλιώς συνεργάζεται μαζί μας ε, τους τελευταίους μήνες, ακριβώς για να εντοπίσουμε και να ε, βρούμε τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε για να περιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο στην καθημερινή δουλειά και να ενσωματώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και όχι μόνο σε αυτό αλλά και στην νόμο παρασκευαστική δουλειά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν κάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις υποβάλλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ένας άλλος εγκάρσιος στόχος και οριζόντιος που έχουμε εντοπίσει εκτός από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι η καλύτερη συνεργασία και η καλύτερη σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική ασφάλεια. Διότι ε, υπάρχει μια τεχνητή ας πούμε διαχωριστική γραμμή ε, ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Μπορεί γι' αυτό να ισχύει κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν υπάρχουν πια σύνορα μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, συνεργασία με τρίτες χώρες, πρώτα με τους εταίρους, τα κράτη-μέλη, αλλά και τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει καλύτερα να είναι ενταγμένο στη στρατηγική μας και πλήρως. Τρίτο στόχος, η καινοτομία. Χρειάζεται περισσότερη δράση πιστεύουμε έτσι ώστε να αξιοποιούμε πλήρως την έρευνα και την καινοτομία και τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν και από την ιδιωτική οικονομία γιατί όχι έτσι ώστε να τα χρησιμοποιούμε αυτά και να μπορούν οι δικαστικές ε, και οι ιδιοκτικές αρχές να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Το τρίτο ε, που ε, βρήκαμε ως εγκάσιο στόχο και κοινό είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά clustering της εσωτερικής ασφάλειας. Τι είναι αυτό. Πρέπει να δημιουργούνται συνέργειες, συνεργασίες μεταξύ της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας και άλλων τομέων πολιτικής. Βεβαίως πάντα αρχής γενομένης από την εξωτερική πολιτική, αλλά θα πρέπει να το συνδέσουμε και με όλες τις άλλες πολιτικές που έχουν επιρροή στην εσωτερική πολιτική ασφαλείας της Ένωσης. Αυτές ε, ας πούμε παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η οικονομία ή οι μεταφορές ή και άλλες πολιτικές που συνδέονται με την ασφάλεια. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσωτερικά αναδιατάσσεται ε, στις υπηρεσίες της για καλύτερη συνεργασία ε, μεταξύ των διαφόρων μονάδων και τμήματων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με θέματα εσωτερικής πολιτικής ασφάλειας. Αλλά για να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στον καθορισμό και στη χάραξη αυτών των πολιτικών. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έχουν κοινό στόχο. Και στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι ακριβώς να ενισχυθεί και ένα συμβουλευτικό φόρουμ ε, το οποίο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λανσάρει στην αυτή στρατηγική έτσι ώστε να ε, συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι φορείς, βεβαίως πάντα οι ε, δημόσιες και κρατικές αρχές που από το ρόλο τους έχουν θεσμική θέση αλλά και οι ιδιώτες και οι πολίτες. Θα αρχίσει αυτό με μια μεγάλη διάσκεψη που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ιταλική Προεδρία να οργανώσει στις 29 Σεπτεμβρίου. 29 Σεπτεμβρίου. Και ε, έχουμε τη χαρά να έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του ο πρόεδρος σας κύριος Μωράες ε, και θα λάβει και το λόγο, αλλά όχι μόνο ο κύριος Μωράες και άλλα μέλη της Επιτροπής σας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν. Ο τίτλος της διάσκεψης, κατά την άποψή μας, δίνει το στίγμα προστασία της κοινωνίας και ε, των δικαιωμάτων των πολιτών με ανανεωμένη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια. Αυτό είναι το έμβριο της μελλοντικής ε, μορφής που θα λάβει αυτή η διάσκεψη που θα είναι ένα συμβουλευτικό φόρουμ γενικότερα τα επόμενα έτη. Αυτά. Κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε θα σταματήσω εδώ να μην μακρηγορήσω. Ε, θέλω όμως να πω ότι η δημόσια διαβούλευση έχει ξεκινήσει ήδη από τις 4 Ιουλίου ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Home και είναι ανοιχτή η διαβούλευση μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Βεβαίως έχουμε καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει και πρόσωπα δηλαδή. Μέχρι τώρα έχουμε μεγάλη ε, ανταπόκριση και επιτυχή. Έχουμε ένα μήνα ακόμα και μέχρι τη διάσκεψη φαντάζομαι θα έχει κορυφωθεί αυτή η προσπάθεια. Θέλω βεβαίως να ακούσουμε και τις δικές σας σκέψεις και απόψεις των αξιότιμων βουλευτών σε σχέση και με το περιεχόμενο της νέας ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Είναι πολλές οι προκλήσεις, χρειάζεται μια κοινή στρατηγική και ελπίζουμε να έχουμε στο πλευρό μας απολύτως το Κοινοβούλιο για να προετοιμάσουμε και τη μελλοντική μας ανακοίνωση που προτίθεται και σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2015. Σταματώ εδώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε, αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να απαντήσω. Να προσπαθήσω τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σορέκα. Έχουμε ορισμένα μέλη που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Κύριος Κύρκοπ. Φαντάζομαι ότι έχετε πληθώρα μελών που θα θελήσουν να λάβουν το λόγο. Ε, είναι ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός ότι η εσωτερική στρατηγική ασφαλείας μας φέρει το ε, ακρόνιμο ISS τη στιγμή που πρόκειται για ακρόνιμο, για παρεμφερές ακρόνιμο μιας μεγάλης τρομοκρατικής οργάνωσης και κράτους. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αλλάξουμε το δικό μας ή να τους, να τους καταστρέψουμε, δηλαδή να τους αφανίσουμε για να μην υφίσταται αυτό το ακρόνιμο πλέον η στρατηγική ασφαλείας μας ε, σαφώς ε, δεν ε, σχετίζεται με τρομοκρατικές απόψεις. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα και θέματα που μας απασχόλησαν ανά το χρόνο που θα πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω και να αναθεωρηθούν ιδιαίτερα ως προς το διεθνές έγκλημα στις κοινέ ομάδες ε, ε, έρευνας. Ήμουν υπεύθυνο λίγα χρόνια πριν ε, σε αυτό το τομέα των κοινών ομάδων αυτών. ξέρω ότι είναι χρήσιμες, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι τις χρησιμοποίησαμε όσο θα έπρεπε. Και με βάση τις διασυνοριακές ε, τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι θα βοηθούσαν ιδιαίτερα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς προχωρούμε σε αυτό το τομέα. Στον ε, τομέα επίσης της τρομοκρατίας, που ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη απειλή, το θέμα, το ζήτημα ενός δικτύου ενσυνειδητότητας, διεθνούς ενσυνειδητότητας και δεν ξέρω κατά πόσο προβλέπεται μια συνεργασία σε αυτό το τομέα μεταξύ κρατών μελών. Ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται δουλειά σε αυτό το τομέα γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ε, τι κίνδυνο διατρέχουν ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε επικίνδυνες περιοχές όπου υπάρχουν σειράξεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πόσο θα προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Επίσης, τι συνεργασία υπάρχει ως προς την επιστροφή ε, πολιτών που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. Ορισμένες ε, χώρες δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτή την επιστροφή πολιτών. Υπάρχει και το θέμα των απάτριδων, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να τους αποδεχτούμε στην κοινωνία μας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σκέφτεστε σε αυτό το τομέα. Τέλος, από τη δική μου άποψη, το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Πάντα βρισκόμαστε πίσω. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τον κυβερνοχώρο και το διαδίκτυο ε, προτρέχοντας ημών. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα σταθούμε στο ύψος των ε, περιστάσεων ή πώς θα ε, εξισορροπήσουμε τις ελευθερίες του κυβερνοχώρου με την πρόληψη του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επίσης, πιστεύω ότι ως προς τη... το... το ζήτημα των ανηλίκων και της βίας κατά των ανηλίκων online, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα της σεξουαλικής ε, κακοποίησης των ανηλίκων και της χρησιμοποίησης τους online είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη σημασία και στα πλαίσια της διαχείρισης του κυβερνοχώρου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να διωχθούν αυτοί που πρέπει, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της ε, χρήσης, της κακής χρήσης των ανηλίκων. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. 7 ε, λεπτά, Αγιάρ. Εντάχει, Λόπες Αγιάρ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσίαση του κυρίου Σορέκα για το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2010 μας απασχόλησε μέσα στα πλαίσια της, της τότε Προεδρίας, μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής στρατηγικής 2010-2014 Εμείς ως Ευρωβουλευτές πώς μπορούμε και πόσο μπορούμε να συνεισφέρουμε μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής ε, στρατηγικής ασφαλείας για τα επερχόμενα χρόνια. Επίσης, η Κομισιόν πώς ε, αποτιμά την κατάσταση, ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Υπάρχει, υφίσταται την έχουμε εξασφαλίσει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. και γραπτός μέσω ψηφισμάτων έχουμε εκφραστεί και έχουμε εντάξει και ορισμένα βασικά ε, ζητήματα μέσα στα πλαίσια της ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παρέμβαση της NSA στην προσωπική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Σορέκα πώς αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα, αυτή η πτυχή της εσωτερικής ασφάλειας. Θα πρέπει να δούμε τη διαφορά μεταξύ εσωτερικής ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, να αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική θεώρηση της μετανάστευσης γιατί συγχέουμε θέματα μετανάστευσης με προκλήσεις εσωτερικής ασφάλειας ή θεωρούμε την ίδια τη μετανάστευση ως πρόκληση στην εσωτερική μας ασφάλεια. Όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής ασφάλειας πώς ε, βελτιώνουμε αυτή την ε, συνειδητοποίηση από τους Ευρωπαίους πολίτες και τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο του όλου θέματος. Και τρίτον, πώς, ε, τι χρήση γίνεται των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων που γίνονται μια φορά το εξάμεινο όπου μιλάμε για την εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθερίες και προσωπική ζωή σε σχέση με, τη, με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Επίσης, όταν συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εσωτερική στρατηγική ασφάλειας για τα επερχόμενα έτη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΛΥΜΠΕ ενέκρινε ένα ψήφισμα σε σχέση με την έρευνα που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, το μεγάλο σκάνδαλο, ως προς το μεγάλο σκάνδαλο ε, υποκλοπών που αφορούσε πρεσβείες, ε, θεσμικά όργανα και ούτω καθεξής. Δηλαδή μπήκαν κοργοί παντού και έγινε μια μεγάλη κατασκοπία κατά των Ευρωπαίων Δημοσίων Υπαλλήλων και θεσμικών οργάνων. Ποια είναι η συνέχεια που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από το έγγραφο αυτό το οποίο θα συζητήσουμε στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο μιλητών γιατί είναι πολλά τα μέλη. Θα διαβάσω τα ονόματα αυτών που είναι ήδη στον κατάλογο και τον κλείνω και σας παρακαλώ θερμά να μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά τώρα. Δύο λεπτά γιατί αλλιώς απαντήσεις δεν θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mrs. Gomez, Mrs. Metzola, Mr. Zdechovsky, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. So if everybody was mentioned, now somebody there. Ποιος είναι εκεί πίσω? Ναι. I close this list now and I give the... Κλείνει ο κατάλογος. Μπόνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, Γενικό Διευθυντή Σορέκα, τον Διευθυντή Σορέκα. Πολύ καλή παρουσίαση και νέες ιδέες. Τρεις ερωτήσεις έχω. Λαμβάνοντας υπόψη τις ε, τραϊκές εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας ε, στην Συρία και στο Ιράκ και την επίθεση του ΙΣΙΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει και με ποιο τρόπο το θέμα των μαχητών ε, στην, ε, που προέρχονται από τις δικές μας χώρες. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό των μαχητών που επιστρέφουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σε, για τα EPA και PNR δεδομένα, σε ποιο σημείο έχετε φτάσει στο διάλογο με τη Ρωσία. Έχει αρχίσει να ισχύει ο νέος κανονισμός Λαμβάνεται υπόψη η τωρινή κατάσταση στην Ουκρανία. Ποια είναι η θέση της Ρωσίας για το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκλειστούν υπερπτήσεις και άλλα μέσα μεταφοράς. Και τρίτον, κάτι που δεν συνδέεται άμεσα με την εσωτερική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων. Ποια συμπεράσματα αντλείτε και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για σας, ε, ποια είναι τα μελλοντικά σας βήματα για αυτή την οδηγία. Νομίζω είναι ζωτική σημασία σε αυτά τα στοιχεία που για την εσωτερική πολιτική. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ τον κύριο Σορόκου. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για την έκθεση εφαρμογής. Εγώ όταν διαβάζω την έκθεση δεν βλέπω μια έκθεση, βλέπω κάποια σαφή σχέδια. Νομίζω όμως ότι χρειαζόμαστε μια έκθεση. Όπως είπε ο κύριος Σκύρκοπ, πού είναι τα τζιτς, πού είναι οι κοινέ ερευνητικέ ομάδες, δεν, δεν, δεν βλέπω τίποτα σχετικό. Και για ποιο λόγο, θέλω να το γνωρίζω. Διότι επανειλημμένα Αποφασίσαμε ότι αυτός είναι ο πυρήνας επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ποια είναι τα αποτελέσματα της στρατηγική μας, πώς έχει εφαρμόστεί. Νομίζω για την κυβερνοασφάλεια ελέγχθη ήδη. Δεν ε, ε, έχουμε συστηματική προσέγγιση για την επιβολή του νόμου στο κυβερνοπεριβάλλον, περιβάλλον, μπορώ να το διατυπώσω έτσι. Κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπουμε καλές ειδες μέσα στην έκθεση. Η δίωξη ατόμων δεν συνιστά συστηματική προσέγγιση, δεν νομίζω ότι επαρκεί. Και κάτι άλλο, πάρα πολύ σημαντικό για μένα, στις 20 Ιουνίου δημοσιεύσατε την έκθεση. Τρεις πριν από τρεις μήνες εξεδόθη σημαντικότατη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μαζική διατήρηση προσωπικών στοιχείων, βάσει της οποίας, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένο λόγος ή συγκεκριμένη υποψία, αντιβαίνει αυτό στο χάρτη ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων άρθρα 7 και 8. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίδραση μέσα στην έκθεσή σας για την πολιτική ασφάλεια για αυτό το ζήτημα. Αναφέρεστε στις ε, επιπτώσεις που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή η απόφαση. Πολύ ωραίο αυτό. Τι εννοείτε όμως, ε, διότι με ζητάτε, εξακολουθείτε να ζητάτε μαζική διατήρηση ε, προσωπικών στοιχείων και ξαναλέω με μαζικό χίδιν τρόπο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και συγκεκριμένη υποψία καλείται και πάλι την ε, να εφαρμοστεί η διάταξη περί διατήρησης προσωπικών στοιχείων. Ποια απάντηση δίνετε εσείς στην απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κέριο το ζήτημα. Πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορείτε απλώς να το αγνοήσετε, θα ήταν σκάνδαλο να αγνοήσετε αυτή την τόσο σημαντική και ξεκάθαρη απόφαση. Ευχαριστούμε Γκόμες. Ε, όχι τόσο για την τωρινή έκθεση, αλλά και για την ε, ανακοίνωση που προετοιμάζεται, για την επικαιροποίηση αυτής της ανακοίνωσης, ήθελα να ρωτήσω το εξής για τους ε, τζιχαδιστές ε, που επανακάμπτουν ε, οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τζιχαντιστές που επιστρέφουν στις χώρες τους. Ποιες προθέσεις έχετε είναι αδιαμφισβήτο ότι συνεργάζονται με εγκληματικές οργανώσεις. Ε, δεν αρκεί λοιπόν η πρόληψη, πρέπει ανά την επιστροφή τους να συλληφθούν και να τους μεταχειριστούμε ε, σαν εγκληματίες. Αλληλένδεται είναι και το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάτι άλλο τώρα. Ε, τι θα γίνει ε, με ε, την επίγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έκρηξη στον επιπολασμό του έμπολα αν φτάσει τελικά στην Ευρώπη Πώς θα συνεργαστούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δράσουν προληπτικά, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα ε, θα μπορούσαμε να το είχαμε προβλέψει πριν από λίγους μήνες και δεν έγινε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναχαιτιστεί ε, η μετάδοση του από τις αρχικές αιστείες. Ε, προσωπικό στους αερολιμένες πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω για την ε, συνεργασία, στην ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Κάποια, κάποιες ένομες τάξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπουν σε περίπτωση διαφθοράς και φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής ε, επιτρέπουν κάποιες συμφωνίες με τους παραβάτες και τέτοιου είδους συμφωνίες ε, εμποδίζουν επιβολή, την επιβολή του νόμου σε άλλα κράτη-μέλη όπως στη Γερμανία παραδείγματος χάρη ε, Πώς θα αντιμετωπίσετε με τέτοια περίπτωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση. Ε, τα μέτρα λιτότητας ε, τρίτων. πώς επηρεάζουν την ε, ικανότητα των κρατών μελών, συγκεκριμένα των κρατών μελών που πλήττονται ιδιαιτέρως από τα, την πολιτική λιτότητας, όπως η χώρα μου, η Πορτογαλία, πώς επηρεάζονται τα κράτη-μέλη ως προς την αντιμετώπιση ε, των ε, μεγάλων σοβαρών απειλών ε, για την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής, παραδείγματος χαρή του ΣΥΕΝΕΡ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μετσόλα, δεν έχουμε διερμηνία στα μαλτέζικα, θα τα πω σύντομα στα αγγλικά. σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ για τους μαχητές θέλω να μιλήσω και για την καταπολέμηση της ρίζος παστικοποίησης βλέπουμε ότι ε, όλο ένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι πηγαίνουν σε εμπόλεμες ζώνες ε, για να συστρατευθούν ε, με τους τζιχαντιστές και μιλάμε για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας που σπρώχνει προς τον εξτρεμισμό. Πολλά κράτη-μέλη μίλησαν για αυξημένες προσπάθειες καταστολής ε, της δράσης αυτών των εξτρεμιστών ε, και έχουμε και το δίκτυο ευαισθητοποίηση για τη ρίζοσπαστικοποίηση και τη σχετική ανακοίνωση του Ιανουαρίου. Βήματα έχουν γίνει για την ριζοσπαστικοποίηση και απορριζοστικοποίηση, ε, όμως πέραν αυτού θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο δράσης μας για να λαμβάνονται ε, υπόψη στοιχεία όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάληψη νέων ε, δράσεων και αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο φαύλο κύκλο μέσα στην ε, πολιτική ασφαλεία, στο νέο ISS. Σας ευχαριστούμε κυρία Ματσόλα, λέει κυρία Γκάλ. Ο κύριος Τσεβνόσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Διευθυντή Σορέκα, σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Άλμπρεχτ. Είναι μάλλον γενικόλογες ε, ως επιτοπλίστων οι παρατηρήσεις Εγώ πάλι έχω ειδικότερα ερωτήματα να σας υποβάλω. Πρώτον, οι μαχητές ε, ε, Τσέχοι, Σλοβάκοι, παραδείγματος χάρη που εμπλέκονται στην σύραξη στην Ουκρανία και εμπλέκονται ε, σε εγκλήματα πολέμου. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εσωτερικών Υποθέσεων έχει κάποια στρατηγική όταν επιστρέψουν, τι σκοπεύει να κάνει προβλέπετε κάποια συντονιστική δράση διεπηρεσιακή στην Επιτροπή. Το καλοκαίρι ασχολήθηκα ε, με το πόσο λειτουργεί η ενισχυμένη βελτιωμένη συνεργασία το, το καλοκαίρι και ε, είδα συγκεκριμένα τη συνεργασία ανάμεσα ε, στις αστυνομικές δυνάμεις της Τσεχίας και άλλες ε, υπηρεσίες. Μπορώ να σας πω λοιπόν πως η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις γερμανικές ε, και τις τσεχικές αστυνομικές δυνάμεις ή τις τσεχικές αρχές επιβολής του νόμου και κολομβιανές ε, αρχές επιβολής του νόμου δείχνουν ότι χρειαζόμαστε 96 ημέρες για να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Αυτά στην εποχή του ίντερνετ. Επανειλημμένα αναφερθήκατε στην καινοτομία. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Μπορείτε ενδεχομένως να μου στείλετε ένα κατάλογο όπου θα απαριθμούνται οι καινοτόμες τεχνολογίες και τα ρηξικέλευθα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί την τελευταία τετραετία. Το περιμένουμε εν υπομονησία το email σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Σορέκα ε, και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, τρεις επισημάνσεις μόνο. Ε, στην περίοδο της κρίσης που διατρέχουν ειδικά κάποιες χώρες του Νότου, ε, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι εθνικές ε, υπηρεσίες, η συνεργασία ε, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Πώς σκοπεύουν να το αντιμετωπίσει αυτό. Διότι η πολιτική, η χάρξη πολιτικής και των μηχανισμών είναι ένα το ζητούμενο, η εφαρμογή τους όμως και από τα κράτη-μέλη είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Σε, αυτή την, ε, στο, σε αυτό ακριβώς το περιεχόμενο και η δεύτερη παρατήρηση που αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Έχουμε δει ότι στις χώρες που διέπονται από μια ε, σκληρή κρίση η περιβαλλοντική ευαισθησία και η εφαρμογή των νόμων σε αυτό το τομέα υποχωρεί. Αν το έχουν παρατηρήσει και αν όντω είναι κάτι το οποίο σκοπεύουν να το αντιμετωπίσουν με κάποια μέτρα. Και το τρίτο, Έχουμε την, ε, και λόγω της ε, κατάστασης στη γειτονιά μας, στην Νότια και την Ανατολική, βλέπουμε ε, ροή προσφύγων η οποία όλο και αυξάνει, ενώ η Ευρώπη κάθεται και συζητάει και προσπαθεί να βρει ε, απαντήσεις σε θεμελιώδη ζητήματα όπως κατηγοροποίηση προσφύγων, όπως ποιος θα παραλάβει ποιους και αν θα τους παραλάβει στο δικό του κράτος ή καλύτερα να πάνε στο γείτονα. Μήπως, έχουμε, ε, μήπως βλέπει και αυτός ότι από τη μία μεριά ε, χτίζουμε αλλά με το άλλο χέρι γκρεμίζουμε γιατί αντί να αντιμετωπίζουμε μόνο το έγκλημα όταν δημιουργηθεί αφήνουμε μια ξενοφοβία, ένα ρατσισμό να διωγγούται και μετά έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ. Σε σχέση με τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τι έκανε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στο παρελθόν έτσι ώστε να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο και όχι απλώς να πληροφορείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ε, δραστηριότητα της προσωρινής Επιτροπής ε, ΚΡΙΜ, ε, η οποία ασχολήθηκε με την διεθνή εγκληματικότητα και ασχοληθήκαμε και με τη μαφία τότε. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο θα πρέπει να επανασυσταθεί η προσωρινή Επιτροπή ΚΡΙΜ και δεύτερον, ποια, ποιο ήταν το έργο και η σημασία αυτής της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης HOME και των εσωτερικών υποθέσεων. Νομίζω το θέμα είναι σημαντικό για την Ιταλία και για την Ευρώπη, διότι η μαφία αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί δικαστές στην Ιταλία απειλούνται, δέχονται απειλές από τη μαφία ως προς τους τζιχαντιστές που ενδεχομένως επιστρέψουν στη χώρα τους. Δεν θα ήθελα να κρατήσουμε την ίδια στάση με αυτή των ε, Αμερικανών. Τη στάση δηλαδή των ΙΠΑ Και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαίοι έχουν παρεκτραπεί λιγάκι ως προς αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να, ξεχ... να ξεχνάμε τις περίφημες renditions στην Ευρώπη, τις παραδόσεις δηλαδή. Και... Ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί πρωτίστως υπόψη. Merci, Madame la Présidente. Κυρία Βεργία. Εμείς όλοι εδώ είμαστε προσιλωμένοι και στην ασφάλεια και την προστασία των πολιτών μας, το δικαίωμα στην ασφάλεια ε, εσωτερική επίσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων όσων διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όμως ότι οι ε, πολιτικές ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών μελών οδηγούν στη λήψη μέτρων που παραβιάζουν και περισσότερο τα δικαιώματα των πολιτών και περιφρονούν μάλιστα και την αρχή της αναλογικότητας. Εδώ είναι τα διάφορα δικαστήρια παίρνουν αποφάσεις. Να σας δώσω δύο θλιβερά παραδείγματα μόνον για ε, την χρήση των προσωπικών δεδομένων και τη μεταναστευτική πολιτική. Είναι μια γάγγρανα αυτή που ε, πλήττει ε, όλο και περισσότερο τα θεσμικά όργανα και μαρτυρία της είναι δυστυχώς η παρούσα ανακοίνωση παρόλο που λέγεται ότι είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής ασφάλειας. δεν θα επαναλάβω τα όσα ακούστηκαν. Ζητώ συγγνώμη για το σκληρό ίσως μου. Δεν μας ενδιαφέρουν εδώ πομφόλιγες και ωραία λόγια, αλλά να κάνουμε πραγματικά μία ε, ανασκόψη, ένα απολογισμό των ε, διαφόρων οργανισμών και του ΙΕ που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και των δικαστηρίων, μίκιο ερευνητές. Ακούσαμε και στην περασμένη θητεία ανησυχίες ε, και αγωνίες, ακόμη και από τον ε, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, σύντομα μία ερώτηση. Πότε θα έχουμε μια ουσιαστική λοιπόν μορφή απολογισμού για το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνέπειες της πολιτικής ασφαλείας στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε τώρα και για ένα συμβουλευτικό φόρουμ. Μπορείτε λίγο να μας ε, εξηγήσετε τι είναι αυτό. Γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε και πάλι με μια μεγάλη δοξολογία, είναι ειδική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά, ε, να κάνει μεγάλες εκδηλώσεις με μικρά, πενιχρά αποτελέσματα. Ε, τέλος, ε, διαβάζουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σιγά σιγά λέει βγαίνουν από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Αυτό που το βρήκατε. Και πού το βασίζεται, διότι όλες οι στατιστικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται να το διαψεύσουν. Αρκεί να δει κανείς μόνο τα στοιχεία της αύξησης της ανεργίας αλλά και της φτώχειας. Ευχαριστώ η κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Διαβάζω στην έκθεση ότι η στατική εσωτερικής ασφάλειας ε, θέλει να προλάβει ε, την ε, τρομοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση. Έχω ερωτήσεις λοιπόν. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσοι είναι υποστηρικτές του Ισλαμικού κράτους και πώς θα το αντιμετωπίσετε, τα έχετε υπόψη σας όλα αυτά. Επίσης, τι γίνεται με τους διαρθρωμένους ελέγχους στα σύνορα. Ε, κυρίως αυτά είναι θέματα εθνικά ε, και η πολιτική ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ιδέουσα. Τι κάνετε για να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με ουσιαστική προστασία των συνόρων για να μην έρχονται στην Ευρώπη υποστηρικτές και οπαδοί του Ισλαμικού κράτους και άλλοι μουσουλμάνοι εξτρεμιστές και τρομοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι τώρα και δίνω το λόγο στον κύριο Σορέκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν πάρα πολλέ ερωτήσει. Είναι πάρα πολύ λίγο ο χρόνο όμω. Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε όσε περισσότερε ερωτήσει μπορείτε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ένα ψήφισμα, είπατε, στη περασμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Τώρα θα συζητήσουν οι συντονιστές τη συνέχεια θα δώσουμε πώς θα παρακολουθούμε και θα πλαισιώνουμε αυτή την προσπάθεια και πώς θα συνεισφέρει η δική μας Επιτροπή στη νέα στρατηγική. Θα το συζητήσουν, επαναλαμβάνω, οι συντονιστές. Ο κύριος Σορέκα, παρακαλώ. Thank you Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της Επιτροπής που έλαβαν το λόγο για να εκφράσουν την άποψή τους και τις ανησυχίες τους. Αυτός είναι και ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να αποφανθεί στην ευρωπαϊκή φιλοδοξία, γενικότερη φιλοδοξία των, της τελευταίας τετραετίας και να εκινήσει μια συζήτηση, όχι να την κλείσει, να την ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει γραπτό ε, κείμενο, η νέα εσωτερική στρατηγική ασφάλειας, για να μην την ε, αποκαλούμε ISS, όπως είπε και ο κύριος Κίρκοπ, θα συνταχθεί το 2015. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας που ξεκίνησε με αυτό το έγγραφο που είναι υπό εξέταση. Και άρα οι απόψεις που ακούσαμε και οι ανησυχίες σας, τα εισαγωγικά σας σχόλια θα συνεισφέρουν στην όλη αξιολόγηση του εγχειρήματος της Κομισιόν. Θα πρέπει να συλλέξουμε αυτές τις απόψεις και να υποβληθούν στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της λίγους μήνες. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. όπως προτίθεστε να κάνετε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όπου όλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Θα έχουμε μια υψηλού επίπεδου συνάντηση στην οποία σας προσκαλούμε και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επανέλθουν για να συζητήσουμε μαζί ως προς τον τρόπο ορισμού μιας ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης αποκλειστικά. Τώρα ως προς ερωτήσεις καθεαυτές Ορισμένες ε, είναι παρεμφερείς, γι' αυτό και θα τις ομαδοποιήσω. Ο κύριος Κίρκοπ αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα και τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν και την διάσκεψη της 29ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή ε, διασυνοριακή τρομοκρατία, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Δύο βουλευτές μιλήσαν για τις ε, κοινέ ομάδες έρευνας ή διερεύνησης. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της τελευταίας πενταετίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υποστήριξαν τις δράσεις της Eurojust, Europol και κρατών μελών. Και η έκθεση αυτή έχει υποβληθεί επίσης. Αλλά θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Συζητάμε το θέμα με τη Europol για να δούμε κατά πόσο σε συνεργασία με τη Eurojust θα προωθηθούν οι δράσεις των κοινών ομάδων έρευνας με την κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη για τα επερχόμενα έτη. Θα επανέλθουμε επί του θέματος. Ως προς τα δίκτυα αυτά ε, τα δίκτυα ε, ρίζωστικοποίησης, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά τα δίκτυα για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία χρήσης των δικτύων από το χρόνο. Ως προς τους ξένους μαχητές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι άκρος ανησυχητικό και σε στενή συνεργασία με το συντονιστή κατά της τρομοκρατίας μέσα στα πλαίσια της ΕΙΕΔ, της δράσης της ΕΙΕΔ. Εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες για τη δράση που θα πρέπει να αναλυφθεί, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο μας έδωσε ε, συγκεκριμένες ενδείξεις κατά την τελευταία του συνάντηση και επίσης το σύστημα πληροφόρησης Schengen έχει τεθεί σε εφαρμογή και τηρείται πλήρως από τα κράτη-μέλη τη στιγμή που αντιμετωπίζουν το θέμα της επιστροφής των ξένων μαχητών. Συμφωνώ με τον κύριο Άλμπρεχτ. ο οποίος ανέφερε ότι η έκθεση είναι πολύ γενική εμβέλειας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι πρόκειται για καταγραφή δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα το οποίο καλύπτει όλες τις εκθέσεις που συντάσσονται από τους επιμέρους οργανισμούς, αλλά και από την Επιτροπή. Μίλησα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, για την ε, δουλεμπορία και για άλλα παρεμφερή ζητήματα. δεν μπορούμε να είμαστε πολύ εκτενείς και φυσικά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι και η μεγαλύτερη πρόκλησή μας εδώ. Πολλά μέλη αναφέρθηκαν στη συλλογή δεδομένων. Η Επιτροπή αυτή από τον Απρίλιο ασχολήθηκε με αυτή την ε, απόφαση του δικαστηρίου για να δει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Η Επίτροπος Μάλστρεμ επέδειξε στεναρή στάση και στην Ολομέλη αλλά και στην Επίτροπή σας και ανέφερε ότι η επόμενη Επιτροπή θα ορίσει τον καλύτερο τρόπο εξισορρόπησης μεταξύ προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας προσωπικών δεδομένων και θεμάτων ασφαλείας. Και γι' αυτό αυτή η έκθεση αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου χωρίς να λαμβάνει θέση όμως επί του θέματος. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε σε συνέργειες και την ανάγκη συντονισμού με άλλες πολιτικές και φυσικά μας βρίσκει πλήρως σύμφωνους. Τα θέματα στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να αποομαδοποιηθούν, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να ορίσουμε την συνολική μας τακτική. Η Γενική Διεύθυνση Home Ζήτησα από όλες τις άλλες υπηρεσίε να συμμετάσχουν σε μία νέα ομάδα αλλά και σε ένα φόρουμ Δεν πρόκειται για κάτι το εντελώς ξεχωριστό, απλώς κάθε χρόνο συλλέγουμε τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συλλέξουν αυτές τις απόψεις και να αλλάξουν αν χρειάζεται την κατεύθυνση της στρατηγικής. Η κυρία Σπινέλη αναφέρθηκε στη δράση της προσωρινής Επιτροπής ΚΡΙΜ. Συμφωνώ ότι η δράση της Επιτροπής ήταν πολύ σημαντική. Εμείς μελλοντικά θεωρούμε ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 25 σημεία του ψηφίσματος 2636 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τα συμπεράσματα της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Γνωρίζω, Πρόεδρε, ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά πρόθεσή μας είναι να επανέλθουμε όποτε το επιθυμείτε για να απαντήσουμε σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σορέκα θα συνεχίσουμε ε, να συνεργαζόμαστε για τα θέματα αυτά και να ε, συζητούμε. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί, που είναι το 6, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών. Το περίφημο PNR ετέθησε ισχύ την 1η Ιουνίου 2012 και τώρα ένα χρόνο μετά ε, γίνεται η πρώτη αξιολόγηση. 29 και 30 Αυγούστου έγινε αυτό το 2013 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει τα βασικά της ευρήματα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Επιτροπή και μετά στην κυρία Νιτβέλτ που ήταν ε, το, η πρώην εισηγήτρια. Παρακαλώ κύριε Σόρεκα, έχετε ξανά το λόγο. Thank you again, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και πάλι να σας παρουσιάσω ε, το αποτέλεσμα της ε, στρατηγικής μας που αξιολογήσαμε πέρσι, τη συμφωνία για το PNR ε, με την Αυστραλία, δείχνει αυτό ότι μπορεί να εφαρμοστεί με καλή διάθεση εκατέρωθεν και να ελέγχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους Αυστραλούς για όλη την άψογη διαδικασία. Όπως είπατε, στην Καμπέρα πέρσι τον Αύγουστο έγινε αυτή η αξιολόγηση μετά το πρώτο έτος εφαρμογής, τον Αύγουστο του 2013. Ήταν εξαμελής η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας εμπειρογνώμων από τις αρχής προστασίας δεδομένων ενός κράτους μέλους. Ήταν η πρώτη λοιπόν, ε, αναθεώρηση. 1η ε, Ιουνίου του 2012 τέθηκε σε ισχύ βασίζεται στο εθνικό δίκαιο της Αυστραλίας που είναι ο νόμος του 88 για την προστασία των δεδομένων και του 1982 επίσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ε, συλλέγονται βάσει της συμφωνίας αυτής. Εκ των προτέρων, ε, μάλλον πριν την αξιολόγησή μας, ε, στείλαμε στο τελωνίο της Αυστραλίας ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο και απάντησαν ε, συμπλήρωσαν οι αρμόδιες ελληνικέ υπηρεσίες και αυτή ήταν ε, ο βασικός μας συνομιλητής κατά τη διάρκεια λοιπόν της ε, αξιολόγησης. Έρχομαι τώρα στο βασικό μας έβριμα. Στο άρθρο 2 της έκθεσης αναφέρεται η γεωγραφική έλλειψη. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις πλέον προς την Αυστραλία. Κάπου πρέπει να σταματήσεις Οπότε 13 ε, είναι οι αερομεταφορείς ε, που ε, ενέχονται σε αυτό με ενδιάμεσους σταθμούς και όχι απευθείας πτήσεις προς την Αυστραλία. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής δεν εντοπίσαμε κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χρήση του PNR για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του σοβαρού και βαριού διασυνοριακού εγκλήματος, καμιά φορά αυτό είναι δύσκολο να οριστεί. Δεν μπορούν να το μετρήσουν αυτό τα δελωνία της Αυστραλίας ε, για το τι συνιστά σοβαρό ή βαρύ διασυνοριακό έγκλημα. Οι αρχές στην Κάμπερα έχουν ε, Ε, πολύ συστηματική προσέγγιση αντιστοίχησης ε, για τα προσωπικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τα PNA, με ηλεκτρονικό τρόπο αφαιρούν και διαγράφουν ε, στοιχεία που είναι πέραν των 19 που αναφέρονται ρητά στη Συμφωνία για τα προσωπικά δεδομένα. Και επίσης σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες της συμφωνίας για τους επιβάτες πάντα, ε, αδιακρίτως εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την ε, εθνικότητα ή τη διαμονή, τον τόπο διαμονής των αλλοδαπών. Την ίδια άποψη έχουν και οι αρμόδιες τελωνιακές αρχές. Ξέρετε ότι απαγορεύεται η διαχείριση και χρησιμοποίηση ευαίσθητων δεδομένων και μας επιβεβαίωσαν οι Αυστραλοί ότι δεν ε, χρησιμοποίησαν ποτέ αυτά τα δεδομένα στην εφαρμογή της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια των δεδομένων, εμείς επαναλαμβάνουμε και επιβεβαιώσαμε ότι έχουν συστήματα και ηλεκτρονικά και ε, φυσικής ασφαλείας. Ε, είναι ε, πάρα πολύ καλά φυλαγμένα, με πολύ περιορισμένη πρόσβαση, ελεγχόμενη για το ποιος έχει ε, πρόσβαση σε αυτό το σύστημα πληροφόρησης. Είναι πάντα κλειδωμένα αυτά τα συστήματα. Ε, είναι διαπιστευμένοι εκείνοι που έχουν πρόσβαση για τον έλεγχο και τα, τα, είχαμε την ευκαιρία να τα διαπιστώσουμε και εμείς αυτά επί τόπου. Ε, σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία. Προβλέπει η συμφωνία ε, ένας αρμόδιος επίτροπος ε, ενημέρωσης στην Αυστραλία να κάνει συχνούς ελέγχους, τακτικούς δηλαδή. Ένας τέτοιος επίσημος έλεγχος έγινε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2012 που έδειξε ότι είναι υψηλό το επίπεδο συμμόρφωσης και επίσης ενημερωθήκαμε ότι αυτό το καιρό διεξάγεται νέα, νέος έλεγχος. Επίσης ο αρμόδιος επίτροπος στην Αυστραλία μας εντυλώσε ότι δεν υπήρχε επιβάτης που να διαμαρτυρήθηκε ή να παραπονέθηκε ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά του δεδομένα ή έτυχαν ε, κατάχρησης. Oh, λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο για την πρόσβαση τώρα. το Τελωνείο της Αυστραλίας έχει λάβει ε, κάποια αιτήματα πρόσβασης, όχι όμως τα προσωπικά δεδομένα PNR. Υπάρχουν και διαδικασίες για να απαντούν εντός 30 ημερών σε τέτοια αιτήματα. Είναι πολύ ε, καλή, εξαιρετική θα έλεγα η εφαρμογή. Και τέλος το άρθρο 13 εξασφαλίζει το δικαίωμα που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ε, να ανατρέχει και να ζητάει και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ε, και ε, γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή η υλοποίηση. Τέλος, το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη μπορεί κάθε φυσικό πρόσωπο να προσφεύγει, είτε είναι ε, παρόν είτε απόν από την Αυστραλία. Υπάρχει ο αντίστοιχο νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, και όταν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση του νόμου μπορεί καθής να ε, προσφύγει. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο όμως. Και τέλος, για την ε, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η λεγόμενη μέθοδος push για την ε, συλλογή αυτών των δεδομένων. Ε, επίσης υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές τις οποίες στηρεί η Αυστραλία. Δύο συστάσεις έκανε η ομάδα μας για να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Η πρώτη σύσταση ήταν ότι θα πρέπει το τελωνίο στην Αυστραλία να τηρεί ε, όσο γίνεται ένα μικρότερο χρονικό διάστημα ε, τα ε, προσωπικά δεδομένα όταν υπάρχει υποψία σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας. Και επίσης θα πρέπει, δεύτερη σύσταση, να μοιράζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση την αναλυτική πληροφόρηση που λαμβάνει η Αυστραλία στα δεδομένα PNR σε συνεργασία με τη Eurojust, τη Europol και τα κράτη-μέλη όταν ζητούν να έχουν τέτοια πληροφόρηση. Το συμπέρασμα της έκθεσης ε, λέγει ότι ε, γενικά η Αυστραλία έχει πλήρως εφαρμόσει ε, τη συμφωνία αυτή βάσει των διατάξεών της και πραγματικά αξιολογούμε πάρα πολύ θετικά και επενούμε την Αυστραλία για αυτή τη στάση ε, και την τήρηση της συμφωνίας βάσει των προδιαγραφών. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας ε, φώτισε η παρουσίαση αυτή. Αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σορέκα για αυτή την ε, λεπτομερή παρουσίαση και δίνω το λόγο στην κυρία Ιντβέλτ που ήταν πρώην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Σορέκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή της έκθεσης αξιολόγησης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της νέας συμφωνίας PNR και την υποστηρίξαμε τη συμφωνία αυτή με την Αυστραλία τότε λέγοντας ότι πρόκειται για έναν ελάχιστο παρονομαστή έκτοτε ε, δυστυχώς έχουμε δεχτεί μια άλλη συμφωνία που δεν αντικατοπτρίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές και αν δω τον κατάλογο άλλων χωρών που ζητούν μεταβίβαση στοιχείων PNR ή εκφράζουν την πρόθεσή τους να κάνουν κάτι τέτοιο, Μεξικό, Ρωσία, Κορέα, Ιαπωνία, τα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική ε, Αραβία και Κατάρ έχουν αρχίσει να συλλέγουν τα στοιχεία από Πέρση, Αργεντινή, Κούβα, Βραζιλία και άλλες ε, προτίθενται να το κάνουν. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και Χαίρομαι, επειδή μας είπε η Επιτροπή ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Για να αρχίσω με τα δύο σημεία επίκρισης. Είπατε ότι τα στοιχεία πρέπει να ε, παρακρατώνται για ε, μία ιδιαίτερα βραχία χρονική περίοδο. Αυτό με ανησυχεί κάπως. Μπορείτε να μου πείτε γιατί οι αρχές της Αυστραλίας ε, παρακρατούν τα στοιχεία για μια πιο μεγάλη περίοδο από αυτή που πραγματικά χρειάζεται. Επίσης, οι πληροφορίες που απορρέουν από το σύστημα θα πρέπει να την χάνουν σωστής αντιμετώπισης ως προς το σε ποιον κοινοποιούνται. Εγώ ως Ολλανδή, αν δω τα τραγικά γεγονότα με το αεροπλάνο ε, το οποίο κατερρύφθη στην Ουκρανία όπου επέβαιναν πολλοί Ολλανδοί και Αυστραλοί, ε, γνωρίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο πληροφόρησης. Μάθαμε επίσης ότι οι Αυστραλιανές αρχές προτίθενται να βελτιώσουν την ακρίβεια των ε, προσωπικών στοιχείων. Αυτό ακούγεται πολύ καλό, αλλά σημαίνει ότι οι αερομεταφορείς είναι αυτοί που θα πρέπει να επιβαρυνθούν με αυτό το κόστος. Γιατί εδώ στη συμφωνία λέμε για τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την όλη ε, εμπορική διαδικασία, δηλαδή οι αερομεταφορείς δεν είναι δημόσιες αρχές, δεν μπορεί να τους ανατεθεί να επαληθεύσουν τα στοιχεία. Θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή κατά πόσο γνωρίζει το πρόγραμμα ε, ακρίβεια στοιχείων ή εξακρίβωση στοιχείων ως προς τη συνεργασία με τις Αυστραλιανές Αρχές. Τέλος, θα γίνει αναθεώρηση της συμφωνίας τέσσερα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ και ε, εδώ θα δούμε πώς έχει εκτελεστεί η συμφωνία από τεχνικής πλευράς και κατά πόσο πραγματικά χρειάζεται αυτή η λήψη και αποθήκευση σωρία στοιχείων. Και ίσως και η οδηγία ε, σε σχέση με την ε, απόρριψη των στοιχείων, δηλαδή τη μη παρακράτησή τους, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εάν σε τρία χρόνια αποτιμηθεί η συμφωνία, τότε η παρακράτηση στοιχείων και η περίοδος παρακράτησης θα ληφθεί υπόψη ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της ε, συλλογής σωρία στοιχείων. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι ε, θα ληφθεί υπόψη το πλαίσιο 360 μέρες μετά τη θέση ισχύ, αλλά πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια σοβαρή αποτίμηση και αξιολόγηση, διότι υπάρχουν στοιχεία που ε, αποδεικνύουν ότι εγκλήματα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη χρήση προσωπικών στοιχείων. Δηλαδή, δικαιολογείται η ύπαρξή τους. Θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν αποφευχθεί εγκλήματα με βάση και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, παρακράτηση στοιχείων. Ο κύριος Κύρκοπ. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και νομίζω ότι ό,τι και να πούμε για τις λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ θετικό που έχουμε την δυνατότητα μιας πλήρους αναθεώρησης, μιας συμφωνίας που έχει τεθεί σε ισχύ. Γιατί υπάρχουν και άλλες συμφωνίες όπως αυτή που εγώ είμαι εισηγητής που αφορούν το PNR και νομίζω ότι οι πληροφορίες είναι χρήσιμες ε, για εμάς. Θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους ότι υπάρχει μία ε, μεγάλη απειλή ε, παγκόσμιας ασφάλειας και έχουμε πέντε χώρες οι οποίες παρακολουθούνται και 14 κράτη-μέλη έχουν τύχη της κατάλληλης χρηματοδότησης για το PNR. Ελπίζω να μην έχουμε μία σωρία συμφωνιών και διατάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε τους κατάλληλους δηλαδή κανονισμούς που να καλύπτουν όλες ε, τις χώρες ως προς τη, τα στοιχεία και τις αφήξεις. Η κυρία Ιντουβέλτ υπέβαλε ερωτήματα ε, ως προς επιμέρους ζητήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες ε, από την Επιτροπή ως προς ε, άλλα στοιχεία που θα ήταν συναφή με μελλοντικές συμφωνίες PNR. Δηλαδή, να αντιλήσουμε τα διδάγματα από το υπάρχον PNR, να είμαστε πιο πειθαρχημένοι και όχι να προβαίνουμε σε τυχές συμφωνίες ε, δεξιά και αριστερά. Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση αυτή δεν, βασι... δεν έγινε από κάποιον ε, δεν συντάχθηκε επί τη βάση των στοιχείων ε, κάποιων που έχουν αρμοδιότητες ερευνητικές είναι μια έκθεση των Αυστραλιανών Αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν αυτό. θα ήθελα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. Σε ποιο βαθμό ε, χρειάζονται είναι απαραίτητα όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απόρριτη. Εγώ πιστεύω ότι δεν αιτιολογείται το να είναι απόρριτη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν χρειάζονται ναι ή όχι όλα τα δεδομένα, διότι αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποια σε δεδομένων τελικά χρειαζόμαστε και να αποτιμήσουμε επακριβέστερα την ε, ανάγκη διατήρησης τη μεταβίβαση των αποθηκευμένων στοιχείων είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε, διότι έχουμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες ε, για τη μεταβίβαση προς τρίτες χώρες, ε, μεταδιαβίβαση ε, προς τρίτες χώρες, και γι' αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν, είναι δεν ανάγκη να κάνουμε διμερείς συμφωνίες. Αν μπορεί εκείνοι να τα μεταδιαβιβάσουν ε, οι Αυστραλιανοί ενώ σε κάποια τρίτη χώρα, τότε δεν θα κάνουν συμφωνίες με μας. Επίσης πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προθεσμίες διατήρησης. Αν άλλη προθεσμία διατήρησης έχει η Αυστραλία και άλλη προθεσμία διατήρησης προβλέπεται μέσα στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει νόημα θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα σημεία και επανέρχομαι και σε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη μέσα στην έκθεση παρότι δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος. Και πάλι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ΕΕ ξεκάθαρα προβλέπει η απόφαση ότι αν δεν ε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο συγγνώμη, κίνδυνος ή η συγκεκριμένη απειλή, συγκεκριμένη υποψία αντιβαίνει στα άρθρα 7 και 8 της Χάρτας ε, των Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, θα το χειριστεί αυτό το ζήτημα. Λέξη δεν λέει γι' αυτό μέσα στην έκθεση. Βάσει αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον βάσει τη κείμενη ενωσιακή νομοθεσία, είναι παράνομα αυτά που κάνουμε. Και γιατί ξέρετε γιατί δεν έχει καταγγείλει κανείς αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν ξέρει κανείς σε ποιον πρέπει να το καταγγείλει. Ε, και μπορώ να προβλέψω και μελλοντική απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουμε να δρούμε ε, παρατυπά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίμπελ ε, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορώ να στηρίξω αυτά που μας είπε η Σοφία Ίντβελντ και ο Γιάνν Φιλίπε Άλμπρεχτ και θα ήθελα ε, να επικεντρωθώ σε δύο σημεία, αλλά πρώτα ε, θα σας έλεγα το εξής, ότι δεν μπορεί δύο να κάνουν το ίδιο πράγμα, απαραίτητα κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Υπάρχουν συμφωνίες που δεν είναι καλύτερες από, αυτές, από τη συμφωνία με την Αυστραλία και σε πολλά σημεία είναι και χειρότερες σε σχέση με την κοινοποίηση στοιχείων προς τρίτες χώρες και άλλα επιμέρους στοιχεία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι με την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, μένουν ανοιχτά πολλά ε, ζητήματα τα οποία δεν συνάδουν με το πνεύμα αυτών που είχαμε θέσει ως στόχους. Αλλά και πάλι θα πρέπει να τονίσω ότι ο αρχικός μας στόχος ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θέλουμε να διωχθεί και να είναι βαριές οι κυρώσεις. Αναρωτιέμαι από πλευράς της Αυστραλίας πόσες ε, στοιχειοθετημένες ε, υποψίες ε, υπήρξαν ε, και στη συνέχεια πόσες κατηγορίες όντως επαγγέλθηκαν επί τη βάση αυτών των υποψιών και τελικά είναι δυνατή μια αποτίμηση σε εφαρμογή αυτών των μέτρων. Δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες δεδομένα έχουν συλλεχθεί. Πού είναι η απόδειξη ότι αυτό επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και το άλλο ζήτημα είναι ότι όταν είναι στοιχειοθετημένη υποψία και πώς στοιχειοθετείται ή όταν απαγγέλλεται μια κατηγορία, ποια ποιες κυρώσεις μιλάμε. Μιλάμε για τις βαρύτερες κυρώσεις που προβλέπονται για τρομοκρατικές πράξεις ε, ή τελικά ε, δεν ε, γίνεται σεβαστό το πνεύμα των αρχικών μας στόχων. Βλέπω ότι και πάλι θα πρέπει να έχουμε μέτρα σύγκριση για να ξέρουμε γιατί ε, πράγμα μιλάμε. Και επανέρχομαι έτσι στο ζήτημα των ε, foreign fighters, ε, των ξένων μαχητών. Γιατί τους ονομάζουμε ξένους αφού είναι Γερμανοί, είναι Άγγλοι, είναι υπήκοοι των δικών μας κρατών, έχουν προσιλητιστεί στο Ισλάμ, έχουν ρίζος παστικοποιηθεί και εμείς τι συζητάμε. Αν θα τους επιτρέψουμε να επιστρέψουν επί τη βάση των κανόνων για το οποίο Συγγνώμη, ε, όταν κάτι πάει στραβά στη χώρα μας, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και... Σίγουρα ε, για να εξασφαλίσουμε την, ε, για να, υπάρχει, να επικρατήσει ασφάλεια στην Ευρώπη για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων σίγουρα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση ακόμη. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε άλλους πέντε συναδέλφους Στίβενς, Γκυγιόμ, Φως, Ένστε και Σπινέλη που έχουν ζητήσει το λόγο και θα κλείσω τώρα τον κατάλογο των ομιλητών διότι 15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Σας παρακαλώ και πάλι να μην υπερβαίνετε το δίλεπτο χρόνο αγόρευσης που σας αναλογεί ώστε να μας μείνουν και λίγα λεπτά για να μας απαντήσει ο κύριος Σορέκα, η κυρία Στίβενς.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 Ε, ερωτήσεις για την Συμφωνία ΕΕ ε, Αυστραλίας. Οι ευαίσθητες πληροφορίες ε, δεν θα διατηρηθούν, δεν θα αποθηκευθούν, μας λέτε. Έχουμε αποδείξεις. Καταρχάς, πώς ορίζουμε την ευαίσθητη πληροφορία. Η θρησκεία, το αν συμμετέχει κάποιος σε ένα συνδικάτο, η φιλετική προέλευση, ποιες είναι οι ευαίσθητες Υπάρχουν φίλτρα, δηλαδή διηθούνται αυτές οι πληροφορίες και διαβιβάζονται. Υπάρχει αυτή η συμφωνία, ωραία, είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας, πολέμηση εγκληματικότητας, πώς γίνεται. Καμιά φορά ε, είναι απαραίτητο να έχει κάποιος ε, στη διάθεσή του και ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, ειδικά στην αντιτρομοκρατική δράση. Έχουμε αυτούς τους μαχητές τώρα που πηγαίνουν στη Συρία. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία μεταξύ αυτών και συχνά υπόσχονται τα κράτη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ουσιαστικά. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή και εύθραυστη αυτή η ισορροπία και πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε και θέλω να μάθω επίσης αν διαβιβάζονται και σε τρίτες χώρες αυτές οι πληροφορίες και αυτό τι σημαίνει, πώς θα χρησιμοποιούν τα κράτη αυτά, ποια κράτη είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον έλεγχο μετά για το πού θα καταλήξουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει κάποια παρακολούθηση, γίνεται, δίνεται συνέχεια. Ε, Υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία. Η Αυστραλία όμω και τα διατηρεί τα στοιχεία και τα διαβιβάζει. Αυτό το κοιτάτε εσείς. Εμείς έχουμε συμφωνία με την Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή φύγουν τα στοιχεία από την Αυστραλία και βρεθούν σε μια τρίτη χώρα. Ποια είναι η μοίρα τους. Εμείς ξέρουμε που πηγαίνουν και τι τα κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την Αυστραλία. Η Αυστραλία ελέγχει και αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιο τρόπο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mrs. Guillaume. Ευχαριστώ κυρία Γκυγιόμ. Εν συντομία, γιατί μιλήσατε για τα δύο λεπτά, ε, η σωστή εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας, ε, τουλάχιστον για τη διατήρηση των στοιχείων έχει μεγάλη ε, σημασία για αυτή τη συμφωνία και για άλλες. Ε, και φυσικά ζωτική σημασία έχει, ε, έχουν οι εγγυήσει που θα έχουμε για την διατήρηση αλλά και για την επαναπροώθηση των στοιχείων σε τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω κάπως την αίσθηση ότι σε αυτή τη θητεία θα ασχοληθούμε πιο εντατικά και θα συζητήσουμε τα θέματα ασφαλείας γιατί από τότε που ε, συνάψαμε και αυτή τη συμφωνία με την Αυστραλία δεν έχει βελτιωθεί ο κόσμος και ο στόχος είναι ε, πάντα ο ίδιος. Όταν έχουμε τρομοκρατία και βαριά εγκληματικότητα και θέλουμε να την ε, αντιμετωπίσουμε δεν ε, μπορούμε να ε, παρακάμψουμε την ανάλυση των δεδομένων ή να την αποφύγουμε. Εντάξει, υπάρχει κάποιο όριο, θα πρέπει να συζητήσουμε μέχρι που φτάνει αυτό, πότε το έχει κανείς ξεπεράσει. Ε, και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και το ΔΕΚ ε, έχει μιλήσει για το θέμα αυτό, πόσο μπορεί κανείς να παρακρατάει τα στοιχεία αυτά, αλλά περνάει η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία, από ό,τι φαίνεται, λειτουργεί καλά Χαίρομαι γι' αυτό και είμαι ικανοποιημένο. Μα λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βαίνει καλώ η συμφωνία. Βεβαίω υπάρχουν και κάποια σημεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή στο μέλλον. Αυτό που είπε ο κύριο Άλμπρεχτ με την ε, περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτε χώρε και η κυρία Νιτφέλ το είπε και για την ακρίβεια των δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει τι γίνεται όταν αυτά ε, δίνονται σε τρίτου. Έχω όμω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα τουλάχιστον σε αυτό το κλάδο ε, θα μας απασχολήσει και ως πρώτο βήμα είναι ένα ελάχιστο ε, μοντέλο, ένα ε, πρότυπο που μπορεί και να εφαρμοστεί και λύσεις να δώσει. Τώρα θα πρέπει ίσως να ασχοληθούμε ε, με κάποια περιφερειακά ζητήματα να τα κοιτάξουμε, τι μπορούμε να προσαρμόσουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία με την Αυστραλία να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Mrs. Ernst. Ευχαριστώ κυρία Ernst. ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι χαιρόμαστε που έχουμε μια τέτοια έκθεση. Δεν αλλάζει όμως τίποτα στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πολύτιμη αυτή και ωφέλιμη συμφωνία. Δεν μας έχετε πείσει. Δεν έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της. Ρωτάω συγκεκριμένα. Πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αποτραπεί. Πόσα αεροπλάνα σωθήκανε από την κατάρριψη. Ε, λίγο πιο συγκεκριμένοι να γίνουμε. Δεν έχω καταλάβει το όφελος αυτής της συμφωνίας. Είναι ένα τέρας τώρα που συλλέγει προσωπικά δεδομένα, ε, που τα συσσωρεύει, χωρίς να υπάρχει πραγματική αιτιολόγηση και πραγματική αξιολόγηση που να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Και παραμένει το ερώτημα, τι τα κάνουν τα δεδομένα πραγματικά, δεν μου απαντάει κανείς αυτό το ερώτημα. Πόσο καιρό τα κρατάνε, πώς τα αναλύουν, πώς τα επεξεργάζονται, σε ποιον τα δίνουν. Αυτά είναι πράγματα που ε, παραμένουν θολά έτσι και σε μια ομιχλώδη κατάσταση που δεν μας βοηθάει. Και αυτό ε, δικαιολογεί και αιτιολογεί την κατάργηση και το ξύλωμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ε, το θεωρώ τυχοδιοκτικό και βάσει και της απόφασης του ΔΕΚ για την διατήρηση των στοιχείων να εκφράζουμε τόσο ικανοποίηση και τόση χαρά για την προληπτική διατήρηση και την απόφαση του ΔΕΚ. Βεβαίως και χρειάζεται μια κριτική ματιά να παρακολουθούμε αυτές τις συμφωνίες και γίνεται και προληπτική ε, ε, ε, παρακράτηση και χρειάζεται μια κριτική αξιολόγηση οπωσδήποτε. Και να πω και κάτι έτσι λίγο κοινικό αν θέλετε. Η Αυστραλία είναι η χώρα ε, από ε, τα πέντε μάτια τα περίφημα που έχουν κάνει τη συμφωνία. Χρειάζεται και PNR με την Αυστραλία. Ε, Θα είμαι πολύ σύντομη. Η Κορνέλια Έρνστ είπε, προείπε αυτά που ήθελα να πω και εγώ, καθώς και η Άλμπρεχτ και Σίπελ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξής. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 30 Αυγούστου, υπάρχει μία ε, σοβαρή σύσταση έτσι ώστε αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία να εγκριθεί το σύντομότερο δυνατόν. Και στη συνέχεια η Επίτροπος Μάλμστρεμ αναφέρθηκε στο ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο παρόμοιων συμφωνιών για την διατήρηση των στοιχείων τουλάχιστον για τους μετανάστες, όπως είπε η κυρία Μάλμστρεμ. Αναρωτιέμαι λοιπόν και υπενθυμίζω αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Άλμπρεχτ. Ε, υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8 η Απριλίου σύμφωνα με την οποία η διατήρηση στοιχείων πέρα μίας περίοδου απαγορεύεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Σορέκα για να μας απαντήσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας δώσω λεπτομερείς πληροφορίες, ξεκινώντας από την κυρία Ιντβέλτ πρώην εισηγήτρια. Την ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία συμφωνία πρότυπο και θα θέλαμε αυτό να αναφερθεί σαφώς ως προς τα δύο σημεία που θίξατε, ως προς τις δικές μας συστάσεις. Όταν είπα ότι καλέσαμε τις Αυστραλιανές Αυστραλιανές ε, τελωνιακές αρχές να διατηρούν αυτά τα στοιχεία ε, μικρό χρονικό διάστημα, αναφέρθηκα στο άρθρο 16 και εκεί όπου πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα μπορούν οι τελωνιακές αρχές να παρακρατήσουν αυτά τα στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όμως ε, προτρέψαμε τις τελωνιακές αρχές να διαγράψουν αυτά τα στοιχεία μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, δηλαδή να μην παρακρατηθούν για πέντε χρόνια, όπως ορίζεται αρχικά. Ως προς την, ε, τις πληροφορίες και την διαβίβασή τους, οργανώσαμε ένα workshop όπου καλέσαμε και εμπειρογνώμονες από την Αυστραλία μαζί με τα κράτη-μέλη τη Europol και τη Eurojust και επετεύχθη συμφωνία με τις τελωνιακές αρχές της Αυστραλίας να μοιράζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Και βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνονται από ανθρώπους που κατανοούν αυτές τις ε, πληροφορίες και στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ λίγες ομάδες ανάλυσης στοιχείων PNR. Άρα μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο ως προς την ακρίβεια στοιχείων. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πρόγραμμα και συνεπώς θα επανέλθουμε επί του σημείου αυτού. Ως προς την αναθεώρηση μετά από μία τριετία δεν θα περιμένουμε την τελευταία στιγμή για να αρχίσουμε την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα και ως προς την περίοδο διατήρηση στοιχείων η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασία της ΙΚΑΟ, η ΙΑΤΑ και WCO και λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πώς εφαρμόζονται αυτές οι πληροφορίες πέρα από την κοινή αναθεώρηση η οποία προβλέπεται. Ως προς την περαιτέρω διαβίβαση, θα ήθελα να επανέλθω στην έκθεση όπου αναφέρουμε ότι οι τελωνιακές αρχές δήλωσαν ότι δεν έχουν διαβιβάσει στοιχεία PNR δυνάμει της συμφωνίας προς τρίτες χώρες. Αυτό αναγράφεται στη σελίδα 16 της συμφωνίας και αναφέρουν ότι γίνονται ανταλλαγές με βάση ε, σχέδια, ταξιδιωτικά σχέδια και με βάση το πρόγραμμα PNR-GOV αλλά καμία ε, πληροφορία δεν έχει διαβιβαστεί σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση διαβίβασης που δεν έχει, δεν έχει γίνει μάλλον δυνάμει της συμφωνίας, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι τα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της συμφωνίας ως προς την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα θα είδατε το παράρτημα Γ της έκθεσης όπου αναφερόμαστε σε περιπτώσεις σοβαρού εγκλήματος ή αντιτρομοκρατίας και ε, σχεδίων που έχουν αποτραπεί εξαιτίας των στοιχείων PNR. Ως προς τα ευαίσθητα στοιχεία, όπως είπε η κυρία Στίβενς, τα ευαίσθητα στοιχεία αποσύρονται και διαγράφονται άμεσα. Και αυτό το αναφέρουμε και στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Σορέκα. Κυρία Ιντβελτ, μισό λεπτάκι σας δίνω. 30 δευτερόλεπτα. Ε, πρώτα απ' όλα... Ε, αυτά που είπατε για τη δεύτερη αναθεώρηση μετά από τέσσερα χρόνια με εξένησαν. Ε, δεν ξέρω τι σχέση έχει με αυτό. Δεν έχει σχέση περισσότερο με αυτό που είπε η κυρία Σίπελ. Να ξέρουμε τελικά είναι ασφαλέστερη η κατάσταση. Και ο κύριος Φως είπε από τότε που εγκρίναμε τη συμφωνία έχει γίνει πιο επικίνδυνος ο κόσμος. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε κάτι πιο σημαντικό για την χρή, από κοινού χρήση των στοιχείων. Εσείς μιλάτε για μονάδες, ε, για τα στοιχεία των επιβατών. Όχι, όχι. Εμείς μιλάμε για ε, ε, δεδομένα που έχουν ήδη αναλυθεί ενδείξεις για συγκεκριμένους κινδύνους οπότε με τις μονάδες επιβολής του νόμου και ασφάλειας πρέπει να έχουμε την αποκοινού χρήση όχι με τις υπηρεσίες που τα συλλέγουν σε επίπεδο επιβατών. Ναι, παρακαλώ. Ε, συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν θέλω να αφήσω αναπάντητο αυτό το ερώτημα της κυρίας Ιντβελ για την περαιτέρα ε, ε αναθεωρησή με ε, η ΚΑΟ και η ΆΤΑ εννοούσα ότι συνεργαζόμαστε με τους Αυστραλούς, τους Καναδούς, τους Αμερικανούς και άλλους και Διαρκώς ε, τους θέτουμε ερωτήματα για να διαπιστώσουμε αν εφαρμόζονται σωστά οι σύμφωνες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ε, αναθεώρησης που γίνεται κάθε 18 μήνες, όχι, κάθε τρίμηνο. Για το δεύτερο σημείο, μάλλον δεν ήμουν ξεκάθαρος. Μα αυτό εννοούσα. Τα ε, δεδομένα προκύπτουν από την ανάλυση για να βελτιωθεί η επιβολή του νόμου στα κράτη-μέλη ε, και η συνεργασία με Europol και Eurojust. Αυτό ζητήσαμε από την Αυστραλία να κάνει, ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστούμε, λέει η κυρία Γκάλ, για τις, ε, την ενημέρωση, για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους ε, για τη συνεργασία τους, για την επικοδομητική τους προσέγγιση. Στις 2.30 θα ξαναέρθουμε και θα συναντηθούμε με την Επίτροπο Μάλμστρομ. Καλή όρεξη.